Okay. Αγαπητοί φίλοι, θα αρχίσω ξανά τη συνεδρίαση. Φορέστε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας γιατί αν μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα δεν θα με καταλάβετε. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλες και όλοι πάλι ξανά στην αίθουσα του ημικυκλίου μετά από το διάλειμμα του καφέ. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, δηλαδή να σχεδιάσουμε τώρα πλέον το τρίτο μέρος της συζήτησης, να συζητήσουμε μέχρι τις 12.30, μία παρά 20 και μετά να ολοκληρώσουμε πλέον την συνάντησή μας. Και θα μας μείνουν λίγα λεπτά για να ακούσουμε την χοροδία. Να παραμείνετε λοιπόν στην αίθουσα ε, λίγα λεπτά. Πάντως δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την μία η ώρα. Έχουμε βέβαια πολλούς ομιλητές εδώ. Ελπίζω να προλάβουμε να τους ακούσουμε όλους και να είσαστε όλοι παρακαλώ σύντομοι. 15 άτομα έχω εδώ και όλοι θα μιλήσουν το πολύ τρία λεπτά. Θα μου άρεσε να είχα και τα ονόματά σας εδώ και τα μικρά σας ονόματα, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό. Γι' αυτό θα σας ε, λέω τον αριθμό της θέσης όπου καθόσαστε. Έτσι λοιπόν είναι πιο εύκολο. Το νούμερο 510. Παρακαλώ.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 Έχετε κάποια ερώτηση. Ήβαν Τόμσον από το Αφροκαραϊβικό Δίκτυο Επιχειρηματιών. Ήμουν στο πρώτο εργαστήριο μέλος. Ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τους εισηγητές που απέδωσαν με πολύ ακριβή τρόπο τα όσα λέχθηκαν στο εργαστήριο. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα ήθελα να πω ακόμη και να δούμε ίσως αν μπορούν να περιληφθούν στο τελικό κείμενο και ιδίως για το να βασιστούμε στην δραστηριότητα της επιχείρησης για να προχωρήσουμε στην οικονομική απελευθέρωση των ατόμων. Είναι σημαντικό κάθε φορά που υποστηρίζουμε οργανώσεις, επιχειρήσεις, αν είναι δυνατό να, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξεκινάνε δικές τους επιχειρήσεις και να τους υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο προσφέροντας την οικονομική ελευθερία, αλλά να μπορέσουν έτσι να αναπτύξουν και τις αστηριότητές τους και τις ίδιες προσωπικότητές τους. Διότι όπου λείπει αυτό, πάλι αυτό είναι ένα είδος φτώχειας. Επομένως η επιχείρηση σαν δρόμος προς την οικονομική αλλά και προσωπική ανάπτυξη. Εκεί θα ήθελα να δω να τονίζετε περισσότερο το θέμα αυτό στα συμπεράσματα. Το άλλο θέμα που ήθελα να σχολιάσω Ένα συνάδελφος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είπε για τα όσα προέκυψαν από το εργαστήρι 3 για την παράγραφο 5 των συζητήσεων όπου η συνάδελφος αυτή είπε να βγάλουμε την ε, λέξη μαύρη Αφρική, το μαύρο αυτό, μαύρη αυτή. Εγώ δεν συμφωνώ. Διότι αυτό υπονοεί ότι ε, δεν υπάρχουν μειονότητες. Αλλά στην ε, Αφρική υπάρχουν 53 διαφορετικές χώρες. Εγώ από τις παρατηρήσεις μου σπάνια βλέπω ε, στα πόστερ και στις διάφορες αφήσει λευκές οικογένειες να βγαίνουν με μικρά παιδάκια και να ζητιανεύουν φαγητό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιληφθεί αυτή η λέξη, αυτό το Black Africa. Το μόνο που νομίζω είναι ότι αυτό το black, το μαύρο Αφρική, δηλαδή πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Θα ζητήσω τώρα το 283 να λάβει το λόγο, που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι μέλος μιας αντιπροσωπείας νέων μια ένωση για τον τρίτο κόσμο. Και θέλω να προσθέσω κάτι που δεν είχα την ευκαιρία να αναφέρω χθε στο εργαστήριο. Η Ευρώπη να δει το ενδεχόμενο να ανοίξει τα σύνορα σε νέους που δεν ανήκουν στην ομάδα έρασμος για ε, ευρωπαϊκές εθελοντικές υπηρεσίες χωρίς δεν είναι υποχρεωτικό να ανοίγει κανείς τον κύκλο έρασμος για τη συμμετοχή στον πολιτισμό μιας άλλης χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολλούς από τους νέους μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπεναράμπ της Ευρωβουλής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι οι περισσότερες παρατηρήσει αφορούν το δικό μας εργαστήριο. Από τη μια μεριά χαίρομαι, από την άλλη μεριά αισθανόμαστε λίγο υπεύθυνοι γιατί δεν καταφέραμε να ενσωματώσουμε όλες τις προτάσεις στο κείμενό μας. Το εργαστήριό μας ήταν πάρα πολύ πλούσιο και αυτό ήταν δύσκολο όλα αυτά να τα συμπτύξουμε σε δύο σελίδες maximum. Μερικές προτάσεις δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης. Στο εργαστήριο υπήρξαν απόψεις διεστάμενες μερικές φορές και ήταν δύσκολο όλα αυτά να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες προτάσεις με ομοφωνία. Επειδή ανήκω στην αριστερά της αριστερά στο Κοινοβουλίου, συγκράτησα λίγο τη γραφίδα μου σε σχέση με ορισμένες προτάσεις, γιατί ως εισηγήτρια φορέας προτάσεων ήθελε οι προτάσεις να είναι συνενετικές και έχει κατά ανάγκη προτάσεις που ενδιαφέρον ιδιαίτερα το δικό μου χώρο. Κάτι άλλο. Οι εργασίες μας κυρίως αναφέρθηκαν παράγγελα με τις εργασίες του εργαστηρίου 1 και ίσως όχι αρκετά στις προκλήσεις για την Ένωση. Ένα σημαντικό που πρέπει να προσθεθεί είναι ότι οι συζητήσει που κάνουμε αλλά δεν υπάρχουν στα στο κείμενό μας είναι η πρόκληση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου όσον αφορά την αντιμετώπιση της φτώχειας. Και ένα δεύτερο στοιχείο πώς θα δώσουμε ζωή στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στη συγκεκριμένη πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου που ήδη υπάρχει και σε προηγούμενα κείμενα είναι ό,τι έχει σχέση με το χάρτη αυτό συν την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ασχολούμαι ειδικά με τα θέματα αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο και πρέπει να δώσουμε και άλλη όθηση. Τρίτο στοιχείο είναι η συζήτηση που είχαμε με διαφορετικές απόψεις στο θέμα Μαύρη Αφρική. και σε μένα και στον Ανδρή θεωρήσαμε σημαντικό αυτή την ιδιομορφία που υφίστανται υπήκοη της, υπήκοοι της ε, Αφρικής κάτω από τη Σαχάρα για να χρησιμοποιήσω αυτό το πιο σωστό όρο ως η κοινότητα, μαύρη κοινότητα που ζει κάπου εμείς θεωρούμε σκόπιμο να παραμείνει η έκφραση αυτή Συμφωνούμε και οι δύο. Εγώ πρότεινα αρχικά πληθυσμό της Βόρειας Αφρικής γιατί θεωρούσα ότι θα έχει περισσότερη ομοφωνία παρά να πούμε κοινότητες Δεν θέλω να επανέλθω σε θέματα που έχουμε πει γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τα σημεία αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε όμως. Τα υπόλοιπα είναι μάλλον λεπτομέρειες. Θα δούμε πώς θα μπορέσουν να μπουν στην τελική εκδοχή του εγγράφου μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ζάγκου Τσάρλι γραπτά έχει ζητήσει το λόγο. Πού είναι. Είναι. Mr. Charlie. Θέλουμε τον κύριο Τσάρλι. Bonjour, Ναι, συγγνώμη, ε, μιλώ εκ μέρου των ε, μαθητών που είναι εδώ. Μιλάτε για τους φτωχούς, για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας περισσότερο. Εμείς όμως που έχουμε εργαστεί με αυτούς τους ανθρώπους, που τους έχουμε δει, που τους έχουμε γνωρίσει, βλέπουμε ότι χρόνια τώρα τίποτα δεν αλλάζει. Όλες αυτές οι προτάσεις που ακούγονται εδώ είναι λόγια του αέρα. Αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται στην καθημερινή του ζωή και δεν τους προσφέρει βοήθεια κανεί και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα υποχρεούνται οι σταξιούχοι να πληρώνουν φόρους. Ενώ όλοι τους στη ζωή δούλευαν και με τους φόρους τους συνέβαλαν στο προϋπολογισμό και άρα τελικά όλες οι προσπάθειές τους πέφτουν στο κενό. Και θα προτιμούσαμε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι συγκεκριμένες, να βλέπουμε κάτι το ορατό και να βλέπουμε μια ουσιαστική αλλαγή. Δηλαδή, λέει ο Πρόεδρος, ας περάσουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει, να, μάλλον ε, υποστηριχθεί συνενετικά από ό,τι φαίνεται. Φριτ, ποιος θα λάβει το λόγο, πού είσαστε. Δεν σας βλέπω, δεν σας βλέπω. Α, εκεί είσαστε, παρακαλώ. Ehm, eh. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω κάτι για την διάσκεψη συνένεση που πρότεινε η διάσκεψη αυτή ακριβώς πριν από τη διακοπή για καφέ. Γιατί ονομάστηκε έτσι η διάσκεψη αυτή συνένεση. Είναι μια συνηθισμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται πολλές φορές σε διάφορες μορφές, αλλά συνήθως είναι 15 άνθρωποι οι οποίοι για δύο μέρες κάθονται και προβληματίζονται πάνω σε κάποια θέματα και καταλήγουν συνενετικά σε προτάσεις. Ως πολίτης όμως της αγοράς, εγώ θα ήθελα να διαφοροποιηθώ από τη συνένεση και να πω ότι δεν είναι δυνατόν η συνένεση να δημοσιευθεί, να βγει προς τα έξω σαν αποτέλεσμα των συζητήσεων ολόκληρης της αγοράς. Γιατί φοβάμαι ότι η μεθοδολογία αυτή δεν έχει να κάνει με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού δεν νομίζω ότι τα αποτελέσματα της διάσκεψης συνένεση δηλαδή μπορούν να θεωρηθούν και τα αποτελέσματα της αγοράς. Από τα διάφορα κείμενα διαπιστώνω ότι υπάρχουν διάφορες τάσεις. Και για μένα υπάρχουν και αρνητικά πράγματα, όπως για παράδειγμα εδώ που λέει ότι δεν υπάρχει σεβασμός για τους μεγάλους και ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται πια για τους ηλικιωμένου. Εγώ θα ήθελα λίγο μεγαλύτερη απόχρωση εδώ, για να μην το πούμε έτσι. Δεν συμφωνώ. Και επειδή συστάσει συστάσεις 1 και δύο, τι αποδείξεις υπάρχουν ότι είναι έτσι. Εγώ δηλαδή σαν πολίτης δεν μπορώ αυτό να το στηρίξω. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να κάνω αυτή την παρέμβαση, αλλά φοβάμαι ότι έπρεπε να την κάνω. Jag vill verkligen understryka att vi ska vara öppna och fria och man har rätt att uttrycka sina åsikter både... Ωραία, νομίζω και εγώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση έτσι κι αλλιώς, οπότε βεβαίως ο καθένας μπορεί να δώσει το... την άποψή του. Ευχαριστώ πολύ. Γαμπριέλα τώρα, εσύ από το κοινωνικό δίκτυο, έχεις το λόγο. Εμένα εννοείται. Ε. Εδώ μπορεί να υπάρχει και άλλη Γαβριέλα, ξέρω. Από την ε, Συμμαχία Εθελοντών για το Ευρωπαϊκό Έτος. Και θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους αυτής της συμμαχίας. Όπως γνωρίζετε το 2011 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Θα ήθελα λοιπόν ιδιαίτερα να εκφράσω τι ευχαριστίε μου για του εθελοντέ που συνεργάζονται στενά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και θέλω να καλέσω όλου εσά και ιδιαίτερα εκείνου οι οποίοι λαμβάνουν τι πολιτικέ αποφάσει για το έτο αυτό το 2011 να δώσετε περισσότερη αναγνώριση σε αυτό το έργο του των εθελοντών μα στην καταπολέμηση τη ένδυα, ιδιαίτερα στι υποδομέ των εθελοντών των εθελοντικών οργανώσεων που αγωνίζονται ε, και που χωρίς αυτές τις οργανώσεις ήταν πολύ χειρότερη κατάσταση για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένδυας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινωνικό αποκλεισμό. Να γίνει λοιπόν η οργάνωση αυτού του έτους ε, με τις, εθελοντικές, τις οργανώσεις των εθελοντών και να στηριχθεί το έργο τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γκαμπριέλα. Όταν ε, αναγυγνώσκω το όνομα κάποιου εδώ στον λόγο, παρακαλώ να σηκώνετε τα, το χέρι σας. Ε, Κασιμίδης, παρακαλώ. Are, you here? Είστε εδώ. Ντόρα, παρακαλώ. Συγγνώμη για το όνομα. My name is Dora Kasimeris. That's why I didn't understand what you said. I'm... <laughs> Ονομάζομαι Dora Κασιμερή και γι' αυτό δεν κατάλαβα τώρα πώς είπατε. Προέρχομαι ε, από την Ελλάδα. Ε, εκπροσωπώ ένα σύλλογο, η Λιαχτίδα, ο οποίος πριν έξι μήνες, οκτώ, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κέντρο φιλοξενίας παιδιού και φιλοξενούμε παιδιά με βαριά νοσήματα από επαρχία, άπορα παιδιά που έρχονται για τα νοσοκομεία των Αθηνών. Ε, μένω σε ένα προάστιο ένα τέταρτο έξω από την Αθήνα και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πρόσβαση πάρα πολύ καλή. Ανήκω στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ το Eurochild και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη χαρά που μου δίνετε να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Το πρόβλημα το μεγάλο και αυτό που δίνει αυτή την ευχαίρεια να μιλήσω είναι η μετανάστευση. Εχθές μάλιστα ανήκω στο, ε, ήμουν στο εργαστήριο 2 είχε πάρα πολύ όμορφη συνεργασία ακούστηκαν απόψεις αλλά δυστυχώς και πολλές αντιδράσεις. Πολύ επικοδομητικές απόψεις Εκεί ήταν μια κοπελίτσα από Βουλγαρία. Ένα κοριτσάκι προσπαθούσε ε, να υπερευσιστεί τη χώρα της. Μάλιστα ήταν δημοσιογράφος όπως δήλωσε και αναφέρθηκε στα σύνορα που προσπαθεί να βάλει η Ελλάδα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα της μετανάστευσης είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή εγώ σαν Ελληνίδα νιώθω ότι ζω σε ένα κήπο με όμορφα λουλούδια, με διάφορα λαχανικά, χωρίς φράχτη. Μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να έχετε ένα όμορφο κήπο και να είναι πανταχώθεν ελεύθερος. Καταλαβαίνετε πώς νιώθουμε. Και εδώ μιλήσαμε για την επίδραση των μεταναστών, μιλήσαμε για την ενσωμάτωση σε μια χώρα που βρίσκεται στα πρόχειρα της φτώχευσης αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, τι να ενσωματώσουμε, τους άστεγους, τους λαθρομετανάστες. Γιατί όταν μιλάμε για μετανάστευση, δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που ήρθαν με τις οικογένειάς τους, εγκαταστάθηκαν, βρήκαν στοργή, βρήκαν δουλειά. Μιλάμε για τους ανθρώπους που περνάνε τα σύνορά μας. Είμαστε παντού σαν ξέφραγο αμπέλι και τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι ανήκουμε στην ίδια κοινότητα. Θα ασχοληθεί ποτέ η κοινότητα με αυτό το πρόβλημα της Ελλάδος ή να έρθω το θέμα της Τουρκίας που καθημερινώς τα αεροπλάνα τους ύπτανται πάνω από την Αθήνα μπορώ να πω, στα όμορφα νησιά μας. Δεν πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Δεν έχουμε όλοι οι Ευρωπαίοι τα ίδια σύνορα. Πού να σταθούμε έχετε αναφέρει σε κείμενά σας τρεις λέξεις την αλληλεγγύη την ευδαιμονία την ασφάλεια ξεχάσατε τη λέξη ανθρωπιά φτάσαμε σε ένα σημείο που χάθηκε από τον έλληνα τον ευαίσθητο η ανθρωπιά. Ζούμε, ε, ζούμε ρατσισμό που δεν τον είχαμε. Όταν πρώτο ήρθαν οι μετανάστες στη χώρα μας τους αγκαλιάσαμε. Αυτή τη στιγμή νιώθουμε εχθρικά. Αυτή απέναντί μας και, μεν, και εμείς απέναντι σε αυτούς. Υπάρχει διαφθορά στη χώρα μας. Ίσως μπορείτε να μου πείτε και ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους τους χρησιμοποίησαν. Ναι, σε πολλά σημεία. Εγώ δεν θα σας πω ότι ζω στη χώρα των αγγέλων, αλλά δεν έχουμε καμιά στήριξη από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Πρέπει κάτι να γίνει. Όλες οι χώρες, Γερμανία, Γαλλία, εσείς εδώ, έχετε σύνορα βάζετε μέσα αυτούς που θέλετε, το νούμερο που θέλετε. Σε εμά μπαίνει ανεξέλεγκτο. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είμαι δύο μέρες στη χώρα σας, είχε καταληφθεί, και δεν ακούω ειδήσει ελληνικές, είχε καταληφθεί η σχολή, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, η νομική από μετανάστες. Μπορείτε να το διανοηθείτε μέσα στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα να υπάρχουν μετανάστες. Δηλαδή, δεν, μπορώ να καταλάβω πού ζω. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω ειλικρινά. Είμαστε απελπισμένοι. Ζω σε ένα προάστιο με 150.000 κόσμο, 10 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και φοβόμαστε μετά τις 8 το βράδυ να βγούμε στο δρόμο. Κι όμως το κοριτσάκι, και δεν το αδικό, ζήτησε, κατέκρινε τα σύνορα, τα τέλος πάντων. Αυτά τα υποτυπώδη σύνορα προσπαθούμε να βάλουμε, να σταματήσουμε αυτή την έλευση των ξένων είναι πολύ δύσκολο. Το πρόβλημα δυστυχώς των χωρών πια δεν είναι μόνο οικονομικό. Το μεγάλο πρόβλημα που, μας διαφθείρει όλους είναι το κοινωνικό. Σκεφτείτε χώρες που μεγαλούν παιδιά χωρίς ανθρωπιά, χωρίς ευαισθησίες. Θα ήθελα αυτό να σας προβληματίσει. Εμείς σαν χώρα πια δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Ζητάμε βοήθεια από εσά και ελπίζω ότι θα την παρέχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο παρακαλώ να λάβει ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της ομάδας συνένεση. Κύριος. Ναι, Πρόεδρε, λαμβάνω το λόγο, διότι φρονώ ότι όσοι έλαβαν μέρος στη έσκεψη συνένεσης στο τέλος αυτό της αγκόρα μπορεί να αισθανθούν πληγωμένοι από τα λόγια που ακούστηκαν εις βάρος του έργου τους. Δεν είναι κανείς ιδιοκτήτης του τίτλου συνένεση ή διάσκεψη για τη συνένεση. Ακόμη και αυτοί που έχουν πολλά χρόνια δουλειά σε αυτήν και τους οποίους και τιμώ. Μόνο η παρακολούθηση, η δουλειά, η προετοιμασία καθιστούν αυτή τη διάσκεψη, διάσκεψη της συνένεσης. Άρα μπορεί κάποια πρόταση που ακούστηκε να μην είχε διατυπωθεί πολύ σκομψά ή να προξενεί επικρίσεις. Αλλά η κάθε πρόταση που έχει προκύψει, προκύπτει ως αποτέλεσμα δουλειάς ανθρώπων που δεν είναι ειδικοί και που μπορεί να μην τα ξέρουν όλα, γιατί αυτό σημαίνει μη ειδικό, αλλά πάντως προσφέρουν τη δική τους εμπειρία και τη δική τους συμβολή σε αυτούς τους χώρους εδώ στις Βρυξέλλες και γι' αυτό θα ήθελα να καταγραφεί όσο μαρτυρία προσωπική και αυθεντική των ανθρώπων που εργάζονται με όσους αντιμετωπίζουν την καθημερινή, τις καθημερινές δυσκολίες της ζωής και νομίζω ότι ως εκ τούτου αυτή η διατύπωση οφείλει, αξίζει τον σεβασμό των άλλων. Hillary Bloom. Hillary, take the Um, microphone. Ένα ή δύο θέματα που θέλω να θίξω. Και λυπάμαι που είμαι η πιο κακότροπη εδώ. Αλλά χρειάζεται θάρρος ακόμα και γι' αυτό. Θα ήθελα παρεμπιπτόντως να αναφέρω κάτι. Γιατί από την ομάδα 1 βλέπω κάτι το οποίο μάλλον εσφαλμένος καταγράφεται ως κανονισμός τραπεζών ήταν κανονισμός δανειοδοτών που δεν καλύπτονται από ρύθμιση. Ενώ οι τράπεζες έχουν, έχουν ενταχθεί σε κανονιστικές ρυθμίσεις. Και επίση θέλω να πω ότι με καταπλήσει αυτή η συνεδρίαση, αν και δεν έχω μεγάλη εμπειρία, δεν πηγαίνω συχνά σε ε, συνεδριάσει γιατί έχω άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Γιατί είναι σαν να προσπαθούμε να μοιήσουμε ανθρώπου ήδη πεπισμένου και μοιημένου. Όλοι μα αγωνιζόμαστε για την αντιμετώπιση τη φτώχεια. Δεν χρειάζεται και πολύ σοφία για να καταλάβει κανεί τι σημαίνει να είναι φτωχό κανεί. Αλλά κάτι το οποίο ξεχνάμε και δεν λαμβάνουμε υπόψη είναι πρώτον ότι έχουμε όλο και περισσότερες δεξιές κυβερνήσεις στις χώρες μας, οι οποίες περιστέλουν την ενίσχυση προς τους φτωχούς και την αρρώγη που προσφέρεται σε αυτούς. Ερχόμαστε εδώ θεωρώντας ότι εμείς είμαστε καλοί, ξέρουμε να φερόμαστε σωστά προς τους φτωχούς και δείχνουν συμπάνη και συμπάθεια και κατανόηση τα προβλήματά τους. Αλλά λησμονούμε ότι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και μάλιστα και οι πλειονότητε των πληθυσμών των κρατών μας, των λαών των κρατών μας, μάλλον δεν συμφωνούν με τα όσα λέμε εμείς. Μάλλον καταφέρονται κατά των φτωχών και θεωρούν ότι ο φτωχός φταίει για τη μοίρα του. Φίρυπιν, όταν μιλάμε για προβλήματα των μεγάλων οικογενειών, πολυτέχνων κτλ. Ε, θα μας πει ο κοινό πολιτή, να μην κάνεις τα παιδιά. Εγώ δεν ακολουθώ αυτό το επιχείρημα, απλώς σας λέγω ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι το προβάλλουν. Και κάτι ακόμη το οποίο δεν ακούστηκε και με καταπλήσει επίσης ότι δεν ακούστηκε είναι ότι δεν ακούστηκε τίποτε για το πόσο υπέτειος μπορεί να είναι κανείς για την ένδυα στην οποία έχει ε, καταπέσει. Και δεν θέλω να ακούγομαι σαν τη Μάρκαρετ Θάτσερ, μακριά από μεν σκέψη, αλλά μην ξεχνάμε τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό. Έχουμε παιδιά, φερρυπίν ναρκωμανών γονιών, εγκαταλελειμμένα, τα οποία μερικέ φορέ μεγαλώνουν οι παππούδε, οι αγιάδε που δεν έχουν και τη δυνατότητα να τα φροντίσουν και να τα προσέξουν όπω πρέπει. Και αυτή είναι μια νέα μορφή φτώχεια αν και δεν είμαι και σίγουρη γιατί αυτή τη μορφή φτώχεια την ε, προξενούσε ανέκαθεν ναι, ο αλκοολισμό. Εν πάση όμω δεν ακούστηκε και θα μπορούσε να συμβάλλει στη συζήτηση το να συζητηθεί το θέμα αυτό. Αντί να λέμε ναι, να κοιτάξουμε τα προβλήματα των γυναικών. Ξέρουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γυναίκε. Και κάτι ακόμη. Άκουσα πολλέ εκκλήσει για περισσότερη έρευνα. Και εγώ λέγω όχι, περισσότερη έρευνα δεν χρειάζεται. Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο λεπτομερή κατανόηση και υψηλέ γνώσει για τα θέματα αυτά. Αλλά βοηθάμε κανέναν με αυτέ τι γνώσει κάναμε από τους φτωχούς. Με αδρά μέτρα, με αδρές κινήσεις μπορούμε να βοηθήσουμε τους κοινούς, τους φτωχούς, χωρίς πολλές λεπτομέρειες και αυτό είναι ακριβώς που χρειάζονται. Και επίσης, όταν ακούω διάφορες ε, αθλειότητες και διαμαρτυρίες ε, για την ε, συνεδρίαση ακούγονται αριθμοί αντί για ονόματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κατάλογο ονομάτων. Αν θέλετε ο κόσμος να αναπτύσσει επαφή μεταξύ του και να αναπτύσσει τη δικτύωση στην οποία αναφερθήκατε, ε, ας μάθουμε τουλάχιστον τα ονόματα ένα του άλλου. Και πώς καταφέρατε να μαζέψετε τόσους λευκούς σε μια συνεδρίαση της Ευρώπης τη σήμερον ημέρα. Πού είναι οι άλλοι, αυτοί που βλέπω εγώ κάθε μέρα στο δρόμο από τις εθνωτικές μειονότητες. Πολύ λίγους βλέπω εδώ. Ε, και αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να, θα πρέπει να το έχετε αντιμετωπίσει. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των ανθρώπων εκείνων που άμεσα, ε, απευθείας δηλαδή εργάζονται στις οργανώσεις βάσης, που εκφράζουν αυτές τις οργανώσεις βάσης, όχι εμάς που αφού κοιτάμε τους φτωχούς από κάποιο θόκο. Και τώρα θα αρχίσω να, γίνω, θα, θα γίνομαι ακόμη πιο δυσάρεστη. Πόσα κόστησε αυτή η συνεδρίαση, κάποιος μου είπε κάπου στα 300.000 ευρώ. Κέρδισε τίποτα κανένα φτωχό από τη συνεδρίασή μα. Δεν νομίζω. Εσεί μπορεί να έχετε μια τέτοια εντύπωση, αλλά πάντω όχι εγώ. Και διερωτώ με, τι του έπιασε αυτού του ανθρώπου να σερβίρουν σαμπάνια σε μια συνεδρίαση για τη φτώχεια. Στον Αβεράνο Βασίλειο, ξέρετε, εμεί την. Την Ευρώπη και αυτούς που δουλεύουν αυτού εδώ τους ε, λέμε συνήθως γουρούνια στο... στο παχνί. Λοιπόν, ήρθα εδώ εγώ ως γουρούνι στο παχνί να με θρέψετε, δεν είχα να φάω. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα κομμάτι ψωμί, ένα μήλο, μια ντομάτα. Το μεσημέρι και το βράδυ πινάκιον φακής. Είναι κανείς φτωχός εδώ ανάμεταξύ μας που έχει ανάγκη να τον ε, ταΐσουμε δωρεάν. Μου προκαλεί αηδία όλη αυτή η κατάσταση. Όταν διαμαρτυρηθήκα, μάλιστα κάποιο είπε: Ε, κάπω έτσι γίνεται πάντα στην Ευρώπη, αυτά είναι τα ευρωπαϊκά στάνταρτ. Μα εγώ δεν θέλω τέτοια στάνταρτ. Δεν θέλω να ζω σαν αυτού του ανθρώπου, ούτε θέλω ο φόρο που έχει πληρώσει και που πληρώνει με τον ΦΠΑ του ο φτωχό άνθρωπο να επιδοτεί τέτοιου είδου συνεδριάσει και οργανώσει ή τμήμα αυτών. Ναυτία μου προκαλούν όλα αυτά. Αντί λοιπόν να τα συζητούμε όλα αυτά, έχω να σα πω τα εξή αυτή την τσάντα που δεν τη χρειαζόμουν και που μου τη δώσατε, την άδειασα. Θα την αφήσω στην πόρτα και παρακαλώ τον κάθε ένα να βάλει από μια πεντάρα για να τη δώσουμε στους φτωχού και στους άστεγους. Γιατί εμείς να έχουμε καλύψει των εξόδων μας τόσο γενναιόδοροι, δεν τη χρειαζόμασταν. Δεν χρειάζεται να βγάλω και κέρδος που ήρθα να μιλήσω σε μια διάσκεψη για τη φτώχεια. Θα αφήνω λοιπόν την τσάντα αυτή εδώ και παρακαλώ τον καθένα να βάλει από μια δεκάρα ό,τι μπορείτε τη συμβολή σα και παρακαλώ την επόμενη φορά προσπαθήστε να είσαστε πιο σωστοί όταν την οργανώνετε. Ευχαριστώ πολύ, Χίλερη. Σε διαβεβαιώνω ότι είχαμε πολλές ισχυρές, θα έλεγα, παρεμβάσεις μέχρι στιγμής και πριν τη δική σου. Συνεχίζουμε με τον Φραντ Βολμάγερ. μετά από την... Εδώ είμαι, Μετά από την παρέμβαση που μόλις ακούσαμε, δύσκολο μου είναι να επανέλθω σε ένα θέμα που νομίζω ότι θύχτηκε αρκετά συχνά στην στο εργαστήρι 1, αλλά δεν εμφανίστηκε τελικά στο τελικό κείμενο για την ε, σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών υγείας που έχουν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση γνωρίζουμε ποιος είναι ο προβληματισμός. Άνθρωποι που χρειάζονται υποστήριξη, άνθρωποι που, έχουν, που προσφεύγουν σε αυτές τις υπηρεσίες γίνονται όλο και περισσότεροι. Αυτές οι υπηρεσίες και τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι είναι και ένας κινητήρας παραγωγής απασχόλησης μέσα σε μια κοινωνία η οποία κατά τα άλλα ασχολείται μονάχα με το κέρδος. Αυτές οι κοινωνικές οι υπηρεσίες λοιπόν ιδρύθηκαν και από ανθρώπους ως μέσα σε μια προσπάθεια αυτοβοήθειας. Αυτές οι υπηρεσίες συχνά αποτελούν μια διασύνδεση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων στην πραγματική, στην καθημερινή ζωή. Πρόκειται δηλαδή για, την, για υπηρεσίες για ανθρώπους ανάπηρους, γέροντες, γυναίκες συχνά, αλλά και επίσης ε, γυναίκες που ε, χρειάζονται απαλλαγή από το φόρτο των οικογενειακών βαρών. Αυτές οι υπηρεσίες συχνά μέχρι τώρα είχαν ένα καθεστώς πάρα πολύ αβέβαιο και πριν από την κρίση. Άρα τα πρόσωπα που εργάζονταν εκεί είχαν αβέβαιη απασχόληση, υψηλό φόρτο εργασίας, κακή αμοιβή. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι οι χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης περικόπτουν πρώτα-πρώτα αυτές συγκεκριμένα τις υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν έχουμε όλο και περισσότερους που χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές, από την άλλη μεριά όλο και λιγότερη χρηματοδότηση, ώστε τελικά επιβαρύνονται οι οικογένειες, επιβαρύνονται οι γυναίκες και επιβαρύνεται και το προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές. Κατατέθηκαν ορισμένες προτάσεις και εγώ θα ήθελα αυτές οι προτάσεις να περιληφθούν στην τελική έκθεση του εργαστηρίου. Πρώτα, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να ψηφιστούν οδηγίες για τις κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικού περιεχομένου, που αυτές να μπορούν δηλαδή τελικά να προσφέρονται με κατάλληλες συνθήκες. Επίσης, αυτές οι υπηρεσίες, είμαι βέβαιος, ότι θα είναι πάρα πολύ ουσιαστική σημασία για ένα κοινωνικό μοντέλο όπως αυτό που επιθυμούμε να δούμε στο μέλλον. Και για μας είναι σημαντικό, αλλά και για τους πολιτικούς είναι σημαντικό να συζητηθεί σε ποιον κόσμο θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν προσφέρουν, συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτού του μοντέλου. Και το τρίτο που έχω να πω είναι να γίνει μια σε βάθος ανάλυση και από πλευρά Ευρωβουλής στις διαπραγματεύσεις που κάνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν δηλαδή, να ασκήσει πίεση ώστε τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων να χρησιμοποιηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας. Ευχαριστώ, Φραντ. Δημήτρης Σταμούλη. Han har Φαίνεται πως δεν είναι παρόν. Κίνγκεν Μπίλεκ. Είμαι εδώ αριστερά σας πρόεδρε. Το 276 την βλέπουμε. Είμαι Πολωνέζα, θα μιλήσω πολωνικά λοιπόν. Είμαι από το Ίδρυμα SOS Life που εξαρτάται από το ε, Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και έχω μερικά θέματα να σας πω σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη της συνένεσης. Ναι, μεν δεν συμμετέχουν εμπειρογνώμονες στο, στη διάσκεψη, ειδική δηλαδή, στη διάσκεψη της ε, συνένεσης. Γι' αυτό το λόγο θέλω να δώσω μερικές προφορίες για τις νέες τεχνολογίες. Αν είναι δυνατό να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες και οι σχετικές συσκευές που ε, χρησιμοποιούνται για αυτές πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν. Έχουν βέβαια ε, οδηγίες χρήσης, αλλά ποιος μπορεί να τις διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Αυτές οι οδηγίες χρήσης είναι φτιαγμένες για επιστήμονες, για ειδικού. Χρειάζεται λοιπόν κάποια γνώση ψυχολογίας και ε, τέτοιων τεχνολογιών. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον κόσμο να κατανοήσει τη γλώσσα των ειδικών προγραμματιστών που φτιάχνουν τα μηχανήματα αυτά. Το άλλο είναι ότι πρέπει να τους δείξουμε, να δείξουμε δηλαδή στους ειδικούς, να σχεδιάσουν τα μηχανήματα αυτά με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανθρώπων. Να μπορούν να χρησιμοποιούνται ενστικτοδός ορισμένα μηχανήματα δηλαδή. Και αφού είναι έτσι και για την επικοινωνία που διευκολύνει τη ζωή μας μέσα στον 21ο αιώνα. Τώρα στο 21ο αιώνα δεν θα πρέπει να χρειαζόμαστε καν τέτοιου είδους οδηγίες χρήσης. Εγώ δεν συμμετείχα σε προηγούμενες διασκέψεις συνένεσης και αυτό που θέλω να σας ζητήσω για το μέλλον είναι, αν μπορείτε, να μας δώσετε συνοπτικά ποιες δράσεις αναλήφθηκαν στη βάση των συστάσεων που έκαναν οι σκέψεις αυτές ή ποιες έρχονται. Δεν έχω ακούσει τίποτε σχετικά. Τι έγινε δηλαδή με τις συστάσεις και τα πορίσματα προηγούμενων διασκέψεων. Γιατί έχω την αίσθηση ότι γίνονται τέτοιες, ε, διεξάγονται τέτοιες ε, συνελεύσεις μόνο σε αυτός σκοπός, μόνο και μόνο για να γίνουν δηλαδή και όχι για να ακουστούν πραγματικά οι γνώμες των πολιτών. Ευχαριστώ. Όλοι μπορούν να πούν τις απόψεις τους. Τώρα όμως δυστυχώς ε, αρχίζει και γίνεται δύσκολο να τους ακούσουμε όλους. Θα σας παρακαλέσω όλους και όλους να είστε σύντομοι. Γιατί αλλιώς σε πέντε λεπτά θα πρέπει να διακόψουμε το γύρο των ερωτήσεων. Εύα Ρόζενμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία παρατήρηση για το εργαστήριο 3. Να αναγνωρίσετε τη σχέση ανάμεσα στην φτώχεια και την πλεονεξία και την αυξημένη κατανάλωση. Γιατί θεωρώ επειδή αναφέρθηκε η λέξη αγγελική αυτό μπορεί να επιτευχθεί η άσκησή της μόνο αν μειωθεί η απληστία, η πλεονεξία και η περιβολική κατανάλωση. Διαφορετικά η αλληλεγγύη θα μείνει κενός λόγο. Οι αξίες της αμοιβαιότητα, της φροντίδας για τους άλλους ε, να πρέπει να υπερισχύσουν του ανταγωνισμού. Πρόεδρος, μου δεν βλέπω το, το επώνυμά σας. Έχετε, έχετε πάντως το λόγο, αν καταλάβατε για ποιον πρόκειται. Ένας κύριος. Okay. About the indicators. Σχετικά με τους δείκτες, στο τρίτο εργαστήριο, δεν ήμουν παρόν γιατί ήμουν σε άλλο εργαστήριο, αναφέρθηκε ότι πρέπει για την καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να γίνουν ετήσιες εκθέσεις απολογισμού με βάση δείκτες. Συμφωνώ. Αλλά θα μπορούσαμε να πάμε πιο πέρα. Ή θα μπορούσαμε να έχουμε γυρίσει και προς τα πίσω. Τι εννοώ. Πολλοί ομιλητές μίλησαν για την άκρη φτώχεια, κίνδυνος για φτώχεια, φτώχεια, Πώς το μετράνε. Άκρα φτώχεια. Σημαίνει απόλυτη φτώχεια. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Οι φτωχοί τι ωφελούνται από τους ορισμούς αυτούς. Αυτό που έχει σημασία είναι η πολιτική που εμείς, οι πολιτικές μάλλον που εμείς θα πρέπει να εγκρίνουμε προκειμένου να καταπολεμηθεί αυτού του είδους η φτώχεια. Τις χρειαζόμαστε. Εγώ ξέρω έναν ορισμό των Ηνωμένων Εθνών. Δύο δολάρια την ημέρα. Αλλά όχι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι το 60% του αντίστοιχου του εξισωμένου εισοδήμου. Πού έχουμε απόλυτη φτώχεια. Έχουμε το όριο του 40% και έχουμε και το 50% το οποίο επίσης και αυτό κυκλοφορεί. Υπάρχουν συγγράμματα που λένε 50-50. Μερικές φορές άλλα λένε 60-40%. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η δική μας κυβέρνηση, όταν μιλάμε για φτώχεια, εμείς λένε «Α, δεν μιλάτε για φτώχεια, μιλάτε για κίνδυνο για φτώχεια, όχι για φτώχεια». Γιατί εδώ μπαίνει αυτός ο όρος «κίνδυνος για φτώχεια» να το βγάλουμε. Μιλήσαμε για έναν δείκτη. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να καταλάβουμε την κατάσταση αν δεν μετρήσουμε και άλλες παραμέτρους. Το, ε, ο, μετρη, ε, ο διαθεσιμότητα που σημαίνει τι λείπει από κάποιον, τι δεν έχει κάποιος, Αν σου λείπουν δέκα, έχεις απόλυτη φτώχεια. Αν σου λείπουν τρία πράγματα, είσαι σε φτώχεια. Η Κομισιόν κάνει μελέτες με στόχο ε, να εισάγει συγκεκριμένε διαδικασίες στον προπολογισμό με έμεσους συλλογισμούς, δηλαδή τι χρειάζεται η μέση οικογένεια, παραδείγματος θα μπει αυτό στη μελέτη της Κομισιόν. Ας ξεκινήσουμε από αυτή τη μελέτη, από αυτούς τους δείκτες. Άλλη μία παρατήρηση για τα πορίσματα των διασκέψεων κονσένσους. Το, το θέμα του βιωτικού επίπεδου Εμείς στο Age Poverty Europe θεωρούμε ότι για τους ηλικιωμένου καλύτερα είναι να υπάρχει ένα καλάθι όσον αφορά το κόστος ζωής που να αφορά ειδικά τους ηλικιωμένους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Μας μένουν maximum 30 λεπτά. Στις μία η ώρα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε σταματήσει. Θα δώσω το λόγο για μερικές αντιδράσεις σε σχόλια από το πάνελ και σε ευρωβουλευτές Αλλάζω λίγο την κατεύθυνση. Λάιλα Γκούρκε, Κόνι Ρόιτερ, Ιζαμπέλ Ντιρό. Πρώτη τελευταία. και άλλος ένας από το πάνελ. Αν περισσέψει χρόνος, θα δώσω το λόγο και στο ακροατήριο, στο ημικύκλιο. Δυστυχώς άλλη λύση δεν έχω, χρονικά. Λάιλα Γκούρκε, πρόεδρος της ε, Κοινωνικής Επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω εδώ σε αυτή την αγορά και να μιλήσω εκ μέρους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ευχαριστώ και την κυρία Ντουνά και τον κύριο Ρούτσεκ. Συγχαρητήρια και στους δυο σας για την οργάνωση της αγοράς αυτής. Νομίζω πως ε, η ουσία που βγήκε είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι αποφασισμένοι να βρουν λύσεις για να υποχωρήσει η φτώχεια από την οποία πλήττονται εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ευθύνη των ε, κρατών μελών. Αυτή είναι μια βασική διάσταση. Οι νέοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βοηθήσει βέβαια να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι εθνικές πολιτικές και θα συνεχίσουμε. Πάντως, μακροπρόθεσμα οι κοινωνικές ε, προκλήσεις έχουν τεράστια σημασία. Υπάρχουν ε, θέματα ήπιες νομοθεσίες όπως είναι ο μη αποκλεισμός, τέτοιου είδους νομοθεσία μπορεί να βοηθήσει τους πολιτικούς να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και τα κράτη-μέλη για το πώς θα προχωρήσουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε τα προβλήματα της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έτσι όπως απορρέουν και από την κρίση. Οι συζητήσεις μας εδώ όμως έδειξαν ότι αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα που αφορούν μόνο τις κυβερνήσεις, αλλά τον καθένα μας, τον κάθε πολίτη χωριστά επίσης. Η μείωση στους εθνικούς προϋπολογισμούς για κοινωνικές υπηρεσίες είναι κάτι που διαπιστώθηκε ακόμα πιο έντονα με την κρίση και αποτελεί απειλή για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αλλά και για τους στόχους της στρατηγικής 2020. Συνεπώς χρειάζεται αμέσως κάποια δράση. Πρέπει να εφαρμόσουμε μια στρατηγική που θα βοηθήσει να συμμετέχουν όλοι στην κοινωνία, να υπάρχει ανελάχιστο ελάχιστο εισόδημα για όλους και πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλους, όπως επίσης και υπηρεσίες ποιότητας για όλους. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι πολιτικές προτεραιότητες φυσικά πρέπει να έχουν και οικονομική στήριξη, γιατί όταν περικόπτονται οι κοινωνικοί προπολογισμοί των διαφορών χωρών, χρειάζεται Απ' την άλλη μεριά κάτι να γίνει για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα στις κοινωνικές μας προτεραιότητες. Η καταπολέμηση λοιπόν της φτώχειας πρέπει να αποτελεί μέρος της οικονομικής μας πολιτικής. Εμείς στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό τα τελευταία χρόνια. Έχουμε φτιάξει μια ειδική ομάδα εργασίας που είχε επαφές ε, και δημιούργησε δίκτυα με οργανώσεις από την κοινωνία των πολιτών και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται συνεργασία που ξεκίνησε την χρονιά την αφιερωμένη στην φτώχεια και συνεχίζεται με ανταλλαγές μεταξύ μας προκειμένου να εκτιμήσουμε τι πρόοδος έχει επιτευχθεί για την επιτευχή των στόχων μας. Επίσης έχουν αναλυφθεί δράσεις προκειμένου να συνειδητοποιήσει περισσότερο ο κόσμος πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα της ένδυας αλλά και πόσο δύσκολε είναι οι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να υπάρξει κάποια αλλαγή. Αν μη τι άλλο, όμω, χρειάζεται η πολιτική βούληση. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ένδια και τα οποία έχουμε εξετάσει φέτο. Εμεί φροντίζουμε για πρωτοβουλίε και εν ώψη τη στρατηγική 2020. Η Ουγγρική Προεδρία από την πλευρά τη έχει ζητήσει διάφορε γνωμοδοτήσει, για παράδειγμα όσον αφορά την οικογενειακή πολιτική και όσον αφορά την κατάσταση των Ρώμα. Θα ξεκινήσουμε και εμείς διάφορες εκθέσεις πρωτοβουλίες που θα ασχολούνται με τους άστεγους, με την κρίση και την εκπαίδευση, αλλά και τη συμπερίληψη των μεταναστών. Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο αλλά και λιγότερο σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει συμμετοχή. Συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική της. Και γι' αυτό η δικιά μας Επιτροπή Οικονομική και Κοινωνική αποτελεί έναν σημαντικό εταίρο και συνομιλητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας προσκάλεσε να έρθουμε εδώ σε αυτή τη τόσο σημαντική συνάντηση της αγοράς που ήταν πιστεύω πετυχημένη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω και προσδοκώ τη συνέχιση της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λέιλα. Θα ήθελα να πω ότι είσαι κάποιος που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα κοινωνικά ζητήματα. Οπότε περιμένω το, τον επόμενο μιλητή τώρα με τη δικιά του εμπειρία. Παρακαλώ. Στέφαν, με πιέζεις ε, πολύ λέγοντας ότι περιμένεις τη συμβολή μας στην κοινωνική πλατφόρμα μπορούμε να συμβάλλουμε στο βαθμό που μα επιτρέπουν οι δυνάμει μα. Θα θέλω να πω ότι είναι μια οργάνωση που δεν ανήκει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι όμω θεσμικό όργανο, διότι αναγνωρίζεται ω εκπροσωπευτικό όργανο των κοινωνικών προσανατολισμού μη κυβερνητικών οργανώσεων και θα θέλω να πω ότι εγώ μπορώ ακόμη και να αναγνωρίσω πολλές ε, την, από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον κοινωνικό τομέα στην Ευρώπη. Τα ονόματά σας τα διαβάζω πολύ γρήγορα, αν τυχόν ξέχασα κάποιον ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά βλέπω με χαρά ότι είστε πολύ εδώ παρόντες και είναι πολύ καλή ευκαιρία που δίνετε. Και άκουσα επίσης, χωρίς να θέλω να πω ότι πρόκειται για λαϊκισμό, κάποιες απόψεις ε, και έκφραση έκπληξη. Σε πάση περιπτώσει όμω θα θέλω να πω ότι καλό είναι να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε στην Ευρώπη. Εγώ ήμουν και στην πρώτη αγορά και στη δεύτερη και με τη νέα νομοθεσία. Ενθυμούμε ότι με το που είχε την ευκαιρία η Ιζαμπέλ να μιλήσει ενώπιον ε, του <laughs> βελγικού ραδιοφώνου είπε εγώ θα αναλάβω την οργάνωση του Αγκόρα και φαντάζομαι και ο κύριο Ρούτσεκ το ίδιο, αν και δεν έχω τόσε γνώσει, έχει εικόνα, να παρακολουθώ το εθνικό του ραδιόφωνο. Η δουλειά μα λοιπόν ποια είναι. Η δουλειά μα είναι να ε, βοηθήσουμε σε μια συνεργατική δράση των θεσμικών οργάνων, όχι να αμφισβητήσουμε την νομοποίηση των Ευρωβουλευτών. Θα ήταν καλό να είχαμε περισσότερου Ευρωβουλευτέ παρόντε, βεβαίω. Και καλό θα ήταν και οι συναδελφοί σα, όχι μόνο εσεί που είστε εδώ, να αναγνωρίσουν ότι έχουν χάσει μια ε, ευκαιρία. Ευκαιρία όχι να μιλήσουν με εμά, γιατί εμά μα βλέπουν κάθε μέρα, συνομιλούμε κάθε μέρα, αλλά να συνομιλήσουν με πολίτε και να καταλάβουν τι ζητάει ο πολίτη και τι ανάγκε έχει. Να κοιτάξουμε τι στατιστικέ. Ο μέσος όρος για τη φτώχεια στην Ευρώπη είναι 40%. 40% μάλλον αυτοί που ψηφίζουν στην Ευρώπη 25% που ε, στο, σε χώρες όπου δεν υπάρχει υποχρέωση ψήφου γιατί ο κόσμος, ο πολίτης δεν βλέπει κανένα λόγο να ψηφίσει. Το 40% λοιπόν το διατηρεί το Βέλγιο που έχει υποχρεωτική την ψήφο, αλλά οι χώρε που δεν έχουν υποχρεωτική τι συμμετοχέ ψηφοφορίε παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Αυτό είναι ένα κακό το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε. Δεν θέλουμε εμεί να κάνουμε τη δουλειά σα, δεν θέλουμε εμεί να μιλήσουμε στο όνομά σα, αλλά πρέπει να καταλάβετε κι εσεί τι είδου δουλειά κάνουμε εμεί, τι είδου έργο επιτελούμε. Χθε και σήμερα στις συζητήσει επίσης ακούστηκε ε, μια αμφισβήτηση του ποιο είναι ο πολιτικό στόχο, λόγο ύπαρξη του Κοινοβουλίου. Κοινωνική πολιτική, κοινωνικέ προδιαγραφέ και όλα αυτά. Πολύ καλά. Ταυτόχρονα μα βλέπουμε ότι είναι μακροσκελή ο κατάλογο, όχι μόνο για την καταπολέμηση τη ένδυα ε, και στην, με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτου, αλλά σε κάθε θέμα που ε, εντάσσεται ζήτημα καταπολέμηση τη ένδυα. Φέρει πίν, κοινωνικέ υπηρεσίε γενικού συμφέροντο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη σχετική έκθεση να ψηφίσει. Εσωτερική αγορά και πράξη την εσωτερική αγορά. Ναι, επίση είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ε, συμφέροντος, με την ενιαία άδεια παραμονής ε, και εργασίας για τους εποχιακούς εργαζομένους. Όλα αυτά πράγματα έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της φτώχειας. Και δεν μπορεί μόνο να ξεχνάμε και την έκθεση Πολυμάτη. Τι σχέση έχει με τη φτώχεια. Ότι ε, πρέπει κανείς να δει από την κρίση τι συμπεράσματα πρέπει να ε, συναχθούν. Ότι η κρίση δηλαδή οφείλεται όχι σε προβλήματα πραγματικά οικονομικά, αλλά στην άκρατη κερδοσκοπία. Αυτή η έκθεση λοιπόν Πολυμάτη μπορεί να δώσει σαφή μηνύματα για τους πολιτικούς σταγούς αλλά και για τον πολίτη. Και δεν θέλω να ξεκαθαρίσω ποια είναι τα σημαντικά για μας θέματα. Αλληλεγγύη καταρχάς. Αλληλεγγύη όχι φιλανθρωπία η, η δική μου η οργάνωση ονομάζεται Solidar και για κάποιο λόγο συγκεκριμένο, γιατί δεν θέλουμε καθόλου φιλαθροπία και λαιμοσύνη. Επίσης γιατί θέλουμε την ανακατανομή των ευθυνών και καλύτερη οργάνωση της αλληλεγγύης μέσα στα κράτη-μέλη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος υπαρξής μας. Δεύτερον, ζήτημα ισότητας. Υπόθηκε ότι ναι, οι ανισότητες ενισχύονται στα κράτη-μέλη, δεν περιορίζονται. Οι πιο φτωχοί γίνονται πιο φτωχοί, οι πιο πλούσιοι πολύ πιο πλούσιοι. Και η μεσαία τάξη συμπιέζεται προς τα κάτω μάλλον, προς την πλευρά των φτωχών. Άρα λοιπόν τι άλλο καινούριο έχουμε εδώ, έχουμε φαινόμενα στα κράτη-μέλη, τους ανθρώπους που έχουν θέση εργασία είναι φτωχοί, δηλαδή δεν αρκεί η δουλειά τους για να τους στρέψει, για να τους εξασφαλίσει τα προστοζήν όλο και λιγότερα κερδίζουν οι άνθρωποι, όλο και πιο πολύ αμφισβητείται η έννοια του κοινωνικού διαλόγου, γιατί δίνονται σε ανεξάρτητους εργολάβους ε, κάποιες δραστηριότητες μιας επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ε, συνεργαστούν, να συνδικαλιστούν οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την ε, φτώχεια και την ένδυα. Έχουμε το άρθρο 9 με την καθοριστική του σημασία, συνθήκη τη ε, Λισαβόνα. Έχουμε τι κοινωνικέ δεσμεύσει στην ε, Ευρώπη του 2020, στον αγώνα για την καταπολέμηση τη ένδυα. Ναι, όλα αυτά μπορεί να μην αρκούν. Όταν όμω φτάνουμε στην θεσμική πλευρά τη δουλειά μα, οπωσδήποτε πρέπει να τα επισημαίνουμε. Ταυτόχρονα έχουμε την οργάνωση ομάδων πιέσεως, ε, ομάδων στρατευμένων, κοινωνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι εδώ παρούσες και μπορεί βέβαια όπως είπατε εσείς να μην είναι μόνο πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών αλλά είναι και πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών και γι' αυτό έχουμε θέση εδώ. Και αυτό ε, σημαίνει ότι έχουμε καθήκον όχι μόνο να προσφέρουμε τη φιλανθρωπία μα και τη βοήθεια σε όποιον την έχει ανάγκη, αλλά να αναλαμβάνουμε και τι ευθύνε μα, να στρέφουμε το βλέμμα και έξω από την Ευρώπη. Τη Βραζιλία, Φερρυπίν, οι κοινωνικέ ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει στη Βραζιλία βοήθησαν τον κόσμο, 20 εκατομμύρια κόσμο να ξεφύγει από τη φτώχεια. Αυτά λοιπόν ξεπερνούν την κλίμακα τη Ευρώπη και νομίζω ότι θα πρέπει να τα συζητήσουμε μέσα στο ορίζοντα των φιλοδοξιών μα. Και πώ μπορούμε συγκεκριμένα να προχωρήσουμε. Τι πρόγραμμα. Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να, ενισχύσουμε, να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης του 2020 και την ε, διελκυστίνδα μεταξύ των ε, δυνάμεων αγοράς και κοινωνικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στα θεσμικά όργανα. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δράσεις πολιτικές, τρόπο καπροσμέτρησης των αποτελεσμάτων τους, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που έχουν άμεση εμπειρία από τη φτώχεια μπορούν ασφαλώ να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια γιατί ξέρουν τι σημαίνει η φτώχεια και τι σημαίνει αποτελεσματική καταπολέμησή τη. Και χρειαζόμαστε και τα μέσα γι' αυτό. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν έχει σαν στόχο μόνο να στηρίζει τα κράτη-μέλη και να του επιτρέπει να ε, αποκρύπτουν ότι δεν ε, κάνουν αρκετέ προσπάθειε για την επαγγελματική κατάρτιση και ότι μόνο ξέρουν να απομίζουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν χρειάζεται το Κοινωνικό Ταμείο να προσφέρει διαρθρωτική ε, στήριξη και ουσιαστική βοήθεια προ του ανθρώπου ώστε να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Πρέπει να δούμε ένα άλλο πρόσωπο τη φτώχεια. Μπορεί να φαίνεται μερικέ φορέ σε συνεδρία όπω σημερινή κάπω δύσκολο, αλλά είναι καλό ότι μπορέσαμε να ακούσουμε για την πραγματική φτώχεια των ανθρώπων που ζουν σε ακρά φτώχεια, σε οικογένειε πολίτεκνε, σε ανθρώπου που ζουν σε, σε απομακρυσμένε περιοχέ και να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο τη φτώχεια, αλλά πολλαπλά. Και αυτό το λέω και για μας, για τα δικά μας τα μέλη, γιατί είναι σημαντικό να δείξουμε όχι μόνο ότι ξέρουμε να δουλεύουμε για τη φτώχεια, ε, αλλά ότι δουλεύουμε και μαζί σας, ότι σας ακούμε, ότι σας βλέπουμε και ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάποιος επέκρινε ότι είμαστε λευκοί. Ναι, παρά είμαστε λευκοί, έχετε δει και σωστή επίκριση, μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό. Άλλο ένα θέμα, αποτελεσματικότητα των πολιτικών στα επίπεδα κρατών μελών. Εμεί στι κοινωνικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει εδώ και καιρό συζητούμε εάν χρειάζονται κοινωνικέ πλατφόρμε στα κράτη-μέλη. Εγώ θα προτιμούσα να οργανωθούν σε όλα τα κράτη-μέλη και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει κοινωνικού προσανατολισμού και να δουν εάν και τα κράτη-μέλη βέβαια μπορούμε να τα πείσουμε ότι υπάρχει ανάγκη για κοινωνικό διάλογο που ίσως δεν είναι πάντα αυτονόητο, αλλά ότι χρειάζεται και συμπληρωματική δράση στον κοινωνικό διάλογο. Αυτό θα βοηθήσει να βελτιωθεί το έργο μας και η αποτελεσματικότητά του. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στον Στέφαν Εσέλ, ένα παιδάρι 93 ετών που πρόσφατα δημοσίευσε στη Γαλλία ένα βιβλίο που τίτλο έχει «Εντινιεβού ντροπή σα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι πραγματικά να αισθανθούμε ντροπή και όνειδος και μετά να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Πριν δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο, έχω να πω το εξή. Βρισκόμαστε εδώ σε μια μεγάλη αίθουσα. Αλλά ταυτόχρονα καθόμαστε και κοντά όλοι μαζί. Βρισκόμαστε σε μια αίθουσα που χρησιμοποιείται μόνο για συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Ευρωβουλής η οποία έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και έκανε μια χειρονομία η Ευρωβουλή απέναντι στην αγορά διαθέτοντάς μας την αίθουσα της Ολομέλειάς της για την διεξαγωγή της συνεδρίασής μας. Για μας είναι σημαντικό ότι μας έδωσαν, μας πρόσφεραν αυτή την αίθουσα και όχι μια οποιαδήποτε. Η Ιζαμπέλ θα λάβει αμέσως τώρα τον λόγο και μας μένουν ακόμα 15 λεπτά. Attendez que j'ai parlé. <laughs> Euh, voilà, donc on... Περιμένετε να μιλήσω πρώτα. Άκουσα πολλά και νομίζω ότι δουλέψαμε πολλά θέματα. Εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο θέλουμε να οργανώσουμε μια αγορά σε τρεις φάσεις. Πρώτον, συμβολή των Ευρωβουλευτών. Είχαμε και σήμερα και χθε στα εργαστήρια. Εμείς οι Ευρωβουλευτές, οι παρόντες, έχουμε ευθύνη να κάνουμε κάτι από αυτά που υπόθηκαν εδώ μέσα. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν ευρωβουλευτέ, να έχουμε μη κυβερνικέ οργανώσει. Πολλοί από αυτέ είστε παρόντε και παρούσε στην αίθουσα και το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο επίσης παρίσταται και τρίτο οι πολίτες οι οποίοι δούλεψαν τις δύο μέρες αυτές πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτή η τριπλή διάρθρωση, κοινωνία των πολιτών, Ευρωκοινοβούλιο, Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο Επιτροπή, μια κοινή προσπάθεια για να μπούμε σε βάθος στα θέματα αυτά. Πολλές προτάσεις γίνανε Μερικές είναι πολύ συγκεκριμένες, παραδείγματος χάρη ε, ειδικό τιμολόγιο για τα κινητά κλπ. Αλλά θέματα και προτάσεις είναι πιο ευραία. Είναι πολλά πράγματα που μας κάνουν να αγανακτούμε. Παραδείγματος χάρη το ότι η οικονομία προέχει της, του κοινωνικού γίγνεσθε. Και άλλε συγκεκριμένε προτάσει που αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο Ευρωκοινοβούλιο για περίφημη στρατηγική του 2020, εγγυημένο εισόδημα κλπ. Άλλε συστάσει ζητάνε να κάνουμε κάτι με μορφή ψηφίσματος που να την ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει πολλά ψηφίσματα καλά και λιγότερο καλά. Αλλά σημασία έχει τι ισχύ θα δώσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα. Έπειτα υπάρχουν ε, προτάσεις που αφορούν άλλου είδους εταίρου. Την ευθύνη, ο κύριο Ρούτσα και εγώ, την ευθύνη μα για την αγορά είναι να πάρουμε όλο αυτό το υλικό, και να στραφούμε πρώτα στη διάσκεψη των Προέδρων, στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου, στους Ευρωβουλευτές της Επιτροπές. Δεν ξέρω με ποια μορφή, πάντως δεσμευόμαστε σε πάγια βάση. Εμείς οι υπεύθυνοι της αγορά θα σας κάνουμε έναν απολογισμό. Να ξέρετε πού κερδίσαμε, πού δεν κερδίσαμε. Γιατί πολλά πράγματα υπόθηκαν εδώ, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσουν ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτε στο Συμβούλιο, και πιθανώ και ούτε και στις χωρέ μέλη. Πάντως δεσμευόμαστε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό, στη σχέση που θα έχουμε μαζί σας. Η κυρία από την Πολωνία ρώτησε η προηγούμενη αγορά τι αποτελέσματα είχε. Η προηγούμενη είχε το θέμα αλλαγή του κλίματος. Θα ξέρετε ότι πριν από τρία χρόνια ήταν κάπως θεωρητικό το θέμα. Σήμερα γίνανε πραγματικά πολιτικό θέμα. Το συζητάει το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, διεθνή βήματα και πολύ σωστά. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα των εργασιών, πάντως έγινε πραγματικό πολιτικό θέμα. Εύχομαι και επιθυμώ το θέμα της άκρας στόχες και της στόχες της στόχες των πληθυντικό θα έλεγα, με όλες τις μορφές της, να γίνει ένα πραγματικό πολιτικό θέμα, όπως έγινε το πρόβλημα για το κλίμα, το ίδιο πράγμα για τη φτώχεια. Να γίνει ένα πραγματικό πολιτικό πρόβλημα για μα, στο Κοινοβούλιο, για την Κομισιόν, για τα κρατημένη και ελπίζω ότι αυτή εδώ η αγορά θα συμβάλλει σε αυτό. Ευχαριστώ. I Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την στράτευσή σας. Βίμπορ Ρούτσεκ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και επίσης όλες και όλους εσάς, είτε πρόκειται για εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, είτε για σας, τις φίλες και φίλους των, ε, της διάσκεψης της συνένεσης, που εδώ αντιπροσωπεύεται τους πολίτες. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε εκλεγμένοι βουλευτές από 27 χώρες και εκπροσωπούμε στο σύνολό μας 500 εκατομμύρια ανθρώπους όπως προσπάθησα να, προσπαθήσαμε να κάνουμε βέβαια τα, τις τελευταίες δύο μέρες ε, κάναμε τις συζητήσεις αλλά γνωρίζουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα ούτε μόνοι της Κομισιόν ούτε μόνο το, το Συμβούλιο των Υπουργών όλοι όπως είπατε και εσείς πρέπει να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα σε όλες τις χώρες και από κάθε πτυχή του ε, θέματος. Δηλαδή και εδώ στο επίπεδο των ευρωπαϊκών οργάνων, θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον, θα ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή, μα ανοίγει τον δρόμο η συνθήκη της Λισαβόνα, συνεργασία δηλαδή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Όπως συστήσατε επίσης πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των χωρών μελών. Διότι ναι, ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα περισσότερα θέματα της ε, κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής παιδείας, ε, αντιμετώπιση της στόχης κτλ. Είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Καμιά φορά μάλιστα η εκπαίδευση σε ορισμένες φορές είναι θέμα αρμοδιότητας των περιφερειών. Πρέπει λοιπόν ξεκινώντας από το ευρωπαϊκό επίπεδο να φτάσουμε μέχρι και το πιο χαμηλό επίπεδο, δηλαδή μέχρι και το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο να ε, βοηθήσουμε να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Και εσείς βέβαια εκπρόσωποι της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών να συμβάλλετε στην προσπάθεια αυτή καθώς επίσης και οι εθελοντές. Άρα δεν είναι σύμπτωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Κομισιόν κήρυξε το 2011 έτος, έτος εθελοντισμού. Είναι περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη που ασχολούνται με εθελοντικέ δραστηριότητε, είτε πρόκειται για τον αθλητισμό, είτε πρόκειται για την παιδεία, είτε πρόκειται για την καταπολέμηση τη φτώχεια, χωρί αμοιβή. Και εμεί εδώ βέβαια ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε μέσα σε όλο τον χρόνο να ενισχύσουμε τι προσπάθειε αυτέ. Ευχαριστώ και πάλι για τις συστάσεις σας. Δεν έχω βέβαια χρόνο για να τις συζητήσω κάθε μια ξεχωριστά. Αλλά όπως είπε η Ελίζαμπετ ήδη, οι συστάσεις αυτές θα διαβιβαστούν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους ηγέτες των ε, κοινοβουλευτικών ομάδων, στους πρόεδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνται με τα οικονομικά θέματα ή με τα κοινωνικά, με την παιδεία, τον πολιτισμό, την ισότητα των φύλων. Η συμβολή σας λοιπόν είναι πολύτιμη. Θα έρθω όμως σε κανένα δυο από αυτές τις συστάσεις. Ευρώπη 2020 είπατε. Και σωστά. Στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμβάλλουμε σε μια πιο συνεκτική δομή για το 2020 που να εγγύψει θέματα στρατηγικής με πιο συντονισμένο τρόπο. Μα συστήσατε επίσης και νομίζω συμφωνούμε όλοι να μην ρίξουμε το βάρος μόνο στα οικονομικά θέματα. Ναι βέβαια, χρειαζόμαστε πιο ξεκάθαρες ε, ρυθμίσεις, χρειαζόμαστε και τους προπολογισμού, αλλά χωρίς να ξεχνάμε τα κοινωνικά θέματα. Και όπως είπατε στις συστάσεις σας, ζούμε στην Ευρώπη έχουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ναι, που διαφέρει καμιά φορά από χώρα μέλος σε χώρα μέλος άρα, αλλά υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα τα οποία μάλιστα έχουν περιληφθεί και στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτά είναι διαφορετικά από αυτά που έχουν οι φίλοι μας στις Ενωμένες Πολιτείες ή στην Ασία. Υπάρχουν και ορισμένες συστάσεις, για παράδειγμα, για το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο ή τα μία. ταμεία. Πάλι και φέτος αλλά και του χρόνου θα συζητήσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2014-2020. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εδώ είναι σημαντικό οι ιδέες σας και οι δικές μας να μπορέσουν να εξοπλιστούν με περισσότερα χρηματοδοτικά κονδύλια. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα ταμεία αυτά, να χρησιμοποιήσουμε και το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο για να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε ορισμένα από αυτά που είπατε για την καταπολέμηση της φτώχειας γιατί όπως είπατε σωστά το επίπεδο της φτώχειας δυστυχώς μέσα στα τελευταία δύο-τρία χρόνια της οικονομικής κρίσης αυξάνεται τα διάφορα επίπεδα της φτώχειας που το συζητήσατε όχι μόνο στο εργαστήρι παριθμών 1 αλλά και στα άλλα. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλες και όλους για τις παρεμβάσεις σας. Δεν πρόκειται να χαθούν, σας το υπόσχομαι και είμαι βέβαιος ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ακούσουν με ενδιαφέρον τα όσα συζητήσατε, τα πορίσματά σας και τώρα ορισμένα πρακτικά θέματα. Ε, ναι, θα τα λάβουμε υπόψη αυτά το θέμα της λίστας συμμετεχόντων για παράδειγμα. Τα σχόλια που κάνατε σχετικά με τι είδους μπουφέ σας προσφέραμε, τα αναψυχτικά κτλ. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Ο αγώνας κατά της φτώχειας δεν είναι εύκολος, το ξέρουμε. Και δεν πρόκειται να κερδιθεί μέσα σε μια νύχτα, αλλά πρέπει να είμαστε επίμονοι και σας υπόσχομαι για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε συνεργασία μαζί σας όχι μόνο για το νομοθετικό μας έργο αλλά και για την διοργάνωση παρόμοιων με την σημερινή εκδηλώσεων. Ναι, θα ήθελα τώρα να σας ευχαριστήσω και εγώ, αγαπητέ Ρίμπορ, καθώς και την Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ στο όνομά σας μάλλον στο πρόσωπό σας ευχαριστώ ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας προσέφερε την θαυμάσια αυτή αίθουσα και χαίρομαι που μπορέσαμε να διεξαγάγουμε εδώ μια τόσο καρποφόρα ε, συνάντηση εγώ εκπροσωπώ την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και δείχνει πόσο καλή είναι η συνεργασία μεταξύ των οργάνων μας. Έχουμε διαφορετικούς ρόλους, αλλά έχουμε και κατά κάποιο τρόπο και ένα κοινό ρόλο, διότι προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για μένα είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι, ανάγκη, ή να αντιληφθούν οι άνθρωποι μάλλον την ανάγκη να υπάρξει μια βιώσιμη Ευρώπη που σημαίνει στην πραγματικότητα μια μακρόχρονη διαρκή ειρήνη. Θυμηθείτε την ευρωπαϊκή ιστορία. Θα ευχαριστήσω και τις και τους διερμηνείς και θα ακούσουμε τώρα την μουσική και ιδίως ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά και το, τα λόγια τραγουδιού θα διαβαστούν. Θα ακούσουμε λίγα λόγια για το κείμενο αυτό, για τα ε, λόγια δηλαδή. Α, μήπως θα μπορούσαν να τα μεταφράσουν οι διερμηνείς. säga Θα συνεχίσουμε στα αγγλικά, δεν χρειάζεται πια να φοράτε τα ακουστικά γιατί στις ε, μία ακριβώς οι διερμηνείς ολοκληρώνουν την εργασία τους, τελειώνει το ωράριό τους άρα δεν θα μεταφραστεί το κείμενο των στίχων του τραγουδιού αλλά ποιος θα το διαβάσει τουλάχιστον. Έχω ένα πλοίο. Ε, το λιμάνι μου είναι δύσκολο. Παραπέω. Ψάχνω ένα βλέμμα. Δώστε μου λίγη ελπίδα. Είμαι μουσικό στο μετρό, από το Μπερσί στο Τροκαντερό. Σε μια μαύρη τρύπα ζω συνέχεια. Ίσως στο τέλος να υπάρχει κάποια ελπίδα. Πουλάω στο πεζοδρόμιο την ψυχή μου και ελπίζω, μόνο ελπίζω. Οι μικροδουλειές, οι άστεγοι, οι μικρές αγγελίες μου δίνουν μια μικρή ελπίδα. Βλέπω το δρόμο μέσα από την τρύπα μου. Σας περιμένω στο διάδρομο που βρίσκομαι να μιλήσουμε λιγάκι, να μου δώσετε λίγη ελπίδα. Έχω ξεκινήσει εδώ και καιρό. Σαν αύτης ήμουν 16 ετών όλη μου τη γνώση θα την έδινα για να μπορέσω να μοιραστώ με κάποιον λίγη ελπίδα. Έχω ένα πλοίο, είναι μια φυλακή και το λιμάνι μου είναι μιζέρια. Παραπέω, ψάχνω ένα βλέμμα, δώστε μου λίγη ελπίδα. Το κείμενο είναι του Λίκ Ζουμπά και η μουσική του Λουίς Μορνέ.